Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε, αλλά περιμένουμε κάποιου συναδέλφου γιατί έχει προβλεφθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Allora, eh, prima di iniziare... Πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, διερμηνείς, ε, οι οποίοι θα διαβάσουν ε, μια ανακοίνωση, παρακαλώ. Ένα μήνυμα από τους διερμηνείς Είμαστε στην 17η ε, μέρα των κινητοποιήσεων ε, και για τις συνθήκες εργασίας ε, και καθότι η δίκηση δεν έχει έρθει σε καμία επαφή μαζί μας για την επίλυση της εργασιακής διαμάχης, σας πληροφορούμε ότι η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώς την προβλεπόμενη ώρα της λήξης της συνεδρίασης. Ευχαριστούμε. Bene, ringraziamo gli interpreti. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους διερμηνείς. Πάμε στο πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης. Προβλέπετε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γι' αυτό σας καλώ να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας κατά τη συνεδρία των συντονιστών χτες, όπως γνωρίζετε αποφασίστηκε να ανατεθεί στην ομάδα EFTD η γνωμοδότηση της πρότασης της Κομισιόν που θέτει το πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον και τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για το πρόγραμμα LIFE. Η ομάδα των σιαλιστών έθεσε αντίρρηση ως προς την απόφαση αυτή την οποία τη βλέπετε στο σημείο 214 των συστάσεων των συντονιστών των πολιτικών ομάδων σας έχουν μοιραστεί χθες Γι' αυτό αποφασίστηκε να ψηφίσουμε για αυτή την αντίρρηση σήμερα το πρωί, έτσι όπως κοινοποιήθηκε από την Γραμματεία της Επιτροπής. Καλείστε λοιπόν τώρα να ψηφίσετε ηλεκτρονικά σε σχέση με την ανάθεση της γνωμοδότησης για το πρόγραμμα LIFE στην ομάδα EFTD. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επομένως, η απόφαση των συντονιστών που ελήφθη χθε μπορεί να προχωρήσει. Τώρα, ο Μαρτίν Χόσλινγκ έχει ζητήσει το λόγο. Χόσλινγκ. Ε, θα ήθελα να εξηγήσω κάτι για τους συναδέλφους που εχθές αποσίασαν. Γιατί γίνεται αυτή η ψηφοφορία τώρα. Πολύ σύντομα. Ε, εχθές τα είπα εκτενέστατα. Είναι πρωτοφανές αυτό που ζούμε. Ως επίτροπή, δίνουμε έκθεση για το κλίμα σε έναν αρνητή της κλιματικής αλλαγής. Το θέμα δεν είναι μόνο το κύρος της Επιτροπής μας, αλλά πώς θα πάμε και στις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Γελιοποιούμαστε πραγματικά. Ξέρω ότι κάποιοι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως ο Άλμπερντες, ε, το βλέπουν ακριβώς όπως και εγώ. στέλνουμε ένα τέτοιον άνθρωπο σοβαρά σε διαπραγματεύσεις. Είναι σκάνδαλο, περίγελος θα έχουμε καταντήσει. Τώρα, φταίνε γι' αυτό το έλκυ φιλελεύθερη, έτσι όπως θα κάναμε, και λυπάμαι πάρα πολύ. Βεβαίως, δεχόμαστε την απόφαση της ε, πλειοψηφίας, αλλά δεν είναι κανό σημάδι για τη μελλοντική συνεργασία μας. Ευχαριστώ, Μάρτιν. Ο Στίβεν έχει ζητήσει το λόγο. Κύριο Άγνιου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι αρνητής του κλίματος. Ξέρω ότι το κλίμα αλλάζει. Όπως γίνεται τα τελευταία 2.000 χρόνια και προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις αλλαγές. Δεν νομίζω όμως ότι η Γεωργία μπορεί να επηρεάσει αυτές τις κλιματικές αλλαγές. Πάντως, εκ μέρου θα έχουμε ένα ευχολόγιο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα θέματα αυτά. Ένα κατάλογο απαιτήσεων προς τους γεωργούς προκειμένου να βελτιωθεί, να αλλάξει ο καιρός παγκοσμίω. Θα ήθελα να εφαρμόσω δύο τεστ αυτές τις ε, ευχές και θα χρησιμοποιήσω την πεντηκοντατή μου πείρα στην, ε, στο, κλάδο αυτό για να εκτιμήσω ε, ποια θα είναι η επίδραση στη γεωργία. Και δεύτερον, ποια θα είναι η επίδραση στο κλίμα. Και θα χρησιμοποιήσω εδώ τις υπηρεσίες από αυτού του Cambridge στην επιστήμη για να αξιολογήσω και αυτό το θέμα. Οπότε θα έχουμε ένα κόστος και ένα αποτέλεσμα. Και πολύ ευχαρίστω ε, να αφισβητήσετε αυτά που θα πω. Θα το προσεγγίσω με την κοινή λογική και την επιστήμη και είστε απόλυτα ελεύθεροι να το αμφισβητήσετε. Συνάδελφοι, δεν είναι τώρα η ώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Για αυτό το σημείο ζήτησε ο Ερίκ το λόγο, θα το δώσω και μετά να περάσουμε στο σημείο 12. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να ζητήσω το λόγο γιατί μίλησε ο κύριος Άγνιο. Απλώς ήθελα να πω ότι η ψηφοφορία αυτή ε, νομίζω θα είναι ιστορική και η σημερινή ημέρα γιατί αρχίζουμε να προετοιμάζουμε την μελλοντική ΚΑΠ 2020-2027 και όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών. Πολλά μέλη της Επιτροπής Άγκρη είναι και στην Επιτροπή Έμβη και ξέρουμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Έμβη, διεκδικεί αποκλειστική αρμοδιότητα για ορισμένα θέματα και επιμερισμένη κοινή συναρμοδιότητα. Οπότε είναι η κατάσταση κάπως ρευστή. Λάθος ήταν η σημερινή ψηφοφορία για να επηρεάσουμε την επόμενη συζήτηση. Γιατί η συζήτηση συνεχίζεται εκκρεμή και δεν μας βοηθάτε καθόλου ούτε τα μέλη της Άγκρη, ούτε τον πρόεδρο Σεκέρσκι να προσπίσουμε τη σημασία της ε, γεωργίας στο κλίμα, στα πλαίσια της προετοιμασίας της μελλοντική ε, ΚΑΠ. Βέβαια, λαμβάνουμε υπόψη και θα δούμε στο μέλλον πώς την ε, συζήτηση που έχει ξεκινήσει ποιος θα βγει κερδισμένος τελικά. Ωραία. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Θα έλεγα τώρα να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Θα πάμε στο σημείο 12, εκεί είχαμε μείνει χθε. Πρόκειται για ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, που αφορά την ανταλλαγή απόψεων για την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κανονισμό που έχει να κάνει με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα ως προς την αξιολόγηση κινδύνου στην διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη που τροποποιεί το γενικό κανονισμό για τα τρόφιμα που υιοθετήθηκε το 2002. Επιπρόσθετα η πρόταση αυτή τροποποιεί οκτώ νομοθετικές πράξεις που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους τομείς της διατροφικής αλυσίδας όπως παραδείγματος χάρη πρόσθεση στις ζωοτροφές, γαματαφόμικρον, ενζήματα, αρωματικές ύλες, υλικά που έρχονται σε επαφή με το τρόφιμα και προϊόντα φυτοπροστασίας και τα νέα τρόφιμα. Η ΕΝΒΗ είναι η αρμόδια επιτροπή, όμως ε, η κυρία Κάντεμπαχ είναι δική μας εισηγήτρια, η φιλοδοξία του Κοινοβουλίου μας είναι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία, σε πρώτη ανάγνωση, προκειμένου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό πριν το τέλος της θητείας μας. Γι' αυτό έχουμε ένα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Επομένως, θα δώσω το λόγο αμέσω στην Κάριν που μπορεί να μας διαφωτίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από πλευρά μου. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από την απόφαση που πήραμε προηγουμένως στην ψηφοφορία, αλλά ας περάσουμε στο θέμα μου. Διαφάνεια και βιωσιμότητα τη εκτίμηση επικίνδυνοτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τροφική αλυσίδα. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ανταλλάξουμε απόψει, τι πρώτε απόψει ακριβώ από την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι πρώτε εντυπώσει να συζητήσουμε. Θέλω να πω καταρχά ότι καλωσορίζω πάρα πολύ την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ταυτόχρονα όμω λυπούμε που ήρθε τόσο αργά η συγκεκριμένη πρόταση. Αν σκεφτούμε ότι εδώ και χρόνια στο Κοινοβούλιο ζητούμε αξιολόγηση ε, της νομοθεσίας ε, της Γενικής για τα Τρόφιμα που εγκρίθηκε το 2002. Να σας πω πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το check-up που κάνουμε, τον έλεγχο. Το 2014-2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτό το REFIT, ε, αξιολογεί και πάλι τη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα. Και ο στόχος αυτού του ελέγχου είναι να δούμε αν ο κανονισμός αυτός εξυπηρετεί ακόμα το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, αν αποδίδει και ε, αν υπάρχει και ε, λογικό κόστος λειτουργίας, πράγμα που ζητούμε και εμείς. Για την γλυφοζάτη, τον Οκτώβριο του 2017 είχαμε την τέταρτη Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία Πολιτών «Σταματήστε τη γλυφοζάτη» και επιδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έθεσε σε κίνηση όλη αυτή την ιστορία για ε, τα φυτοφάρμακα και τις διάφορες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου. Το Δεκέμβρη του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα οδικό χάρτη για την πρόταση αυτή σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα και μέσα σε τέσσερις εβδομάδε, αντί για τι 12 που ε, είναι η κανονική προθεσμία, έπρεπε να γνωμοδοτήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Πέσαν και τα Χριστούγεννα και δεν είχε και τεράστια πύχη αυτή η διαβούλευση. 20 μόνο ε, ενδιαφερόμενοι απάντησαν. Στι 15 Γενάρη ολοκληρώθηκε αυτό το check-up και παρουσίασε το αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΔΕ Απρίλιο έκανε τη νομοθετική πρόταση. Τα αποτελέσματα αυτού του check-up τι δείχνουν, ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, διαφάνεια σε ό,τι αφορά την εκτίμηση κινδύνου σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία. Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, δηλαδή να μην χωνεύουμε, να μην, να μην ε, ε, δεχόμαστε ε, αυτά τα στοιχεία που θεωρεί η βιομηχανία απόρριτα, να είναι και απόρριτα, αλλά θα πρέπει να δημοσιεύονται. Ε, όταν κάποιο καταθέτει αίτηση για να διοδοτηθεί ένα προϊόν ή μια ουσία θα πρέπει να δικαιολογεί το απόρριτο και να δηλώνει ξεχωριστά ποια στοιχεία θεωρεί απόρριτα. Όταν υπάρχει υπόνοια για κίνδυνο της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων του περιβάλλοντος, θα πρέπει να δημοσιεύονται και όλες οι απόρριτες ε, πληροφορίες θα πρέπει στην ιστοσελίδα του ΕΦΣΑ οι μελέτες να είναι ε, αναρτημένες σε ένα σημείο εύκολο για τον αναγνώστη να το βρει και για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Τώρα, Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα, πνευματικά δικαιώματα, πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία μπορούν να επικαλεστούν ε, εκείνοι που ζητούν άδεια κυκλοφορίας. Ε, αυτά ισχύουν ήδη για κάποιες ουσίες που δεν ε, δημοσιεύονται. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό επιστημονικών μελετών ε, και η ΕΦΣΑ να τα ανακοινώνει αυτά νωρίς για σκοπούς διαφάνειας και δεν μπορεί να χρησιμοποιούν και να επικαλούνται μόνο μελέτες που συνηγορούν υπέρ της έγκρισης κυκλοφορίας μιας ουσίας. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με εκείνους που επιλέγουν εργαστήρια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουν τις επιστημονικές μελέτες. Γενικώ ε, διαβουλεύσεις, δημοσιεύσεις, ε, ανακοινώσεις ε, για τα συμφέροντα, για τις μελέτες που σχεδιάζονται σε περίπτωση αναθεώρηση ή ανανέωσης της άδεια μιας ουσίας που έχει ήδη εγκριθεί. Όλα αυτά αυξάνουν τη ε, διαφάνεια και ανταποκρίνονται στι απαιτήσει. Θα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσο τα εργαστήρια ε, τηρούν ε, τι προδιαγραφέ και οι μελέτε γίνονται με σωστό τρόπο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου, θα πρέπει ο Οργανισμό για την Ασφάλεια Τροφίμων να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται οι μελέτες και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, αποτελεσματικότερη ενημέρωση για το σύνολο των κινδύνων. Ε, μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερη ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε μία διετία ε, θα πρέπει να εγκρίνει ένα γενικό σχέδιο για την ε, ανακοίνωση των κινδύνων και με εξουσιοδότηση πράξης δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού. Εγώ αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό νομοθέτημα το θέμα της πληροφόρηση και δεν πρέπει να είναι αντικείμενο κάτι εξοδό της Πρέπει να την ξαναδούμε την πρόταση. Ε, αλλαγές στη διοίκηση του οργανισμού ΕΦΣΑ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη. Επίσης θα υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα φροντίζει οι επιστήμονες να είναι πολιτικά και οικονομικά ανεξάρτητοι και να υποστηρίζονται και να χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά από την ΕΦΣΑ για να ενισχύει την επιστημονική συνεργασία. Έτσι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διορίζει ή να προτείνει πολλούς εμπειρογνώμονες. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ε, πτυχές της νομοθετικής πρότασης και όπως σας είπα με τις δικές μας τροπολογίες θα λάβουμε υπόψη πολλά θέματα δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Στόχος μας είναι η αύξηση της αξιοπιστίας της ΕΦΣΑ στην ανάλυση κινδύνου και η δημιουργία του σχετικού νομικού πλαισίου. Αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε ε, μόνο εφόσον αυξηθούν οι πόροι του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων και οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί για να μπορούν να κάνουν και δικές τους μελέτες εσωτερικές. Πολλές καλές ιδέες έχουμε καταρχήν, οι οποίες όμως χρειάζονται ακόμα επεξεργασία ε, έτσι ώστε να ε, έχουν επιτυχή ε, εφαρμογή. Σας είπα ότι υπάρχει τρομερή πίεση χρόνου και προσβλέπω στη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την εντολή για τον τριμερή διάλογο ακόμα στην παρούσα θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Κάριν για την παρουσίαση. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμερα έχουμε εκπρόσωπο της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ, θα δώσω το λόγο στην αδελφο Σράιερ. 29-30 Αυγούστου να υπενθυμίσω ότι θα εξετάσουμε ε, το σχέδιο της γνωμοδότησης, προθεσμία για τις τροπολογίες 5 ε, Σεπτεμβρίου και έγκριση της γνωμοδότησης 22 Οκτωβρίου. Ε, κυρία Σχράια, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ. Πρώτον, υποστηρίζω το στόχο τη πρόταση για μεγαλύτερη διαφάνεια για την αξιολόγηση κινδύνου, για βελτίωση τη ποιότητα και τη ανεξαρτησία των επιστημονικών μελετών και την καλή λειτουργία του οργανισμού ΕΦΣΑ. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει συγκεκριμένη πρόταση ε, για να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του check-up του ελέγχου της νομοθεσίας. Έχω όμως τέσσερα ερωτήματα. Πρώτον, δημόσιο μητρό επιστημονικών μελετών. Είναι καλό στις προθέσεις ε, αυτή η πρόταση, αλλά υπάρχει εμπιστευτική πληροφόρηση που πρέπει να προστατεύεται. Και δεν θα πρέπει να τα αποφασίζει αυτό ο οργανισμός ΕΦΣΑ. Θα πρέπει το σύστημα να παραμείνει αποτελεσματικό, γιατί πολλοί ανησυχούν για το Μητρό αυτό που θα είναι δημόσιο, μήπως προκύψει επιπλέον διοικητικό κόστος και για τον ΕΦΣΑ και για τις επιχειρήσεις και θα χάσουμε το αποτέλεσμα και το στόχο μας. Και ε, προβληματίζονται οι επιχειρήσεις. Δεύτερον, βελτίωση της ποιότητας και της ανεξαρτησίας των επιστημονικών μελετών με επιπλέον βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας σε ελέγχους, σε εργαστήρια και δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητάει επιστημονικές μελέτες ίδια. Ωραία όλα αυτά. Ε, ε, έγκαιρη ενημέρωση στον ΕΦΣΑ με στάνταρ τρόπο και ένα σύστημα πληροφόρηση, δημοσίευση, βέβαια με εμπιστευτικότητα. Όλα αυτά είναι θετικά. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε και τα ανεξάρτητα επιστημονικά εργαστήρια για την ασφάλεια τροφίμων πραγματικά πρέπει να είναι στο προσκήνιο και είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι ε, μεθοδικοί και ανεξάρτητοι οι επιστήμονες. Τρίτον, συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΑ των κρατών μελών. Συμμετέχει λοιπόν ένα από κάθε κράτος μέλος, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, ο κλάδος και η ΜΚΟ. Έχω μια παρατήρηση να κάνω ανανέωση του πάνελ μετά από μία πενταετία και διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και πρόληψη κινδύνου. Τολμώ να το αμφισβητήσω. οι επιστήμονε όταν είναι συνδεδεμένοι επί μία πενταετία με το πάνελ αυτό που θα παραμείνουν ανεξάρτητοι και πώς ε, θα βελτιωθεί η λειτουργία. Τέταρτο, καθόλου ευκαταφρόνικο, το, η ενημέρωση για τον κίνδυνο. Στην Ολλανδία αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, προβλέπει ένα τέτοιο σχέδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό είναι αυτό. Πρόσφατα είχαμε Ε, στην κρίση του Φιπρονίλ εσφαλμένη ενημέρωση από τους αρμοδίους στην Ολλανδία και αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ενημέρωση που θα πρέπει να γίνεται σωστά για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και για την ασφάλεια της πληροφόρησης ε, των πολιτών που θέλουν ε, υγιεινά τρόφιμα. Δεν θα πρέπει να διαδίδονται διάφορες φήμες Τα πάνελ της ΕΦΣΑ έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη λειτουργία και την ενημέρωση. Και για πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να συνεδριάζουν για να ε, έχουμε οικονομία χρόνου και χρήματος. Μπορεί να γίνει με τρόπο πιο σύντομο και πιο αποτελεσματικό. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει επίση να γίνονται οπωσδήποτε και έλεγχοι. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριο Χάουσλινγκ έχει ζητήσει το λόγο. Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Χτες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Επίτροπο για το θέμα αυτό. Γενικά η πρωτοβουλία μου αρέσει και θα την υποστηρίξουμε. Κλείνει το μικρόφωνο. Υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε εκτενώς. Δηλαδή, μέχρι πού θα φτάσει τελικά η διαφάνεια, ποια είναι τα εμπορικά απόρριτα. Πολλές επιχειρήσεις θα πούνε ότι αυτό είναι μυστικό, είναι εμπορικό, ε, απόρριτο και προστατεύεται. Και το συζητήσαμε και με τον Επίτροπο και διμερός. Και το ρώτησα αυτό μέχρι πού φτάνει σε επίπεδο εταιρεία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η έδρα τους πώς μπορείς να υποχρεώσεις τρίτους να τηρούν τους κανόνες. Και κάτι που έχει αποφασιστική σημασία είναι η ενίσχυση του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΦΣΑ. Είδαμε ότι έχουμε προβλήματα να βρούμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονε. Τα κράτη-μέλη δεν στέλνουν ανεξάρτητους εμπειρογνώμονε στα πάνελ του ΕΦΣΑ για διάφορου λόγου. και μεταξύ άλλων ε, ότι δεν έχει λεφτά ο οργανισμός και θα πρέπει να κάνει τώρα και ανεξάρτητους ελέγχους θα πρέπει να έχει ε, το απαραίτητο δυναμικό και πόρους για να θέτει αυτές τις ανεξάρτητες μελέτες. Γενικώ καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή και υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ελπίζω να ξεκαθαριστούν για να αποφασίσουμε στην παρούσα ακόμη θητεία, διότι πρόκειται και για την ίδια την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και τα τελευταία χρόνια έχει στραπατσαριστεί αυτή και θα πρέπει να τη επανορθώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρτιν. Σουσάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Παόλο. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η νομοθεσία αυτή και θα μας βοηθήσει να ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε και πάλι τη λειτουργία μας. Να πω κάτι που είπε και ο Μάρτιν Χόισλενγκ τώρα μόλις και θέλω να το υπογραμμίσω κι εγώ γιατί είμαι υπέρ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους θεσμούς που έχουμε ήδη και τα όργανα που έχουν αυτή την αποστολή. Να κάνω μία σύγκριση. Κοιτάξτε τον ΕΟΦ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έμα. Έχει και το θεωρώ σε αυτό το διπλάσιο προϋπολογισμό και το διπλάσιο προσωπικό από την ΕΦΣΑ. Και, και χαίρομαι γι' αυτό, δεν λέω ότι δεν χρειάζεται, αλλά περισσότερα τρόφιμα παίρνουμε παρά φάρμακα, έτσι δεν είναι. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε ε, να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του αυτός ο οργανισμός, να φροντίζει για τη διαφάνεια και τη σωστή ενημέρωση και να συνεχίσουν να κυκλοφορούν καλά τρόφιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σουζάννα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ε, εδώ είναι ο κύριος Μπόχορτ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΑ Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Είμαι ευγνώμων για τα πολύ θετικά και θαρρυντικά σχόλια και την υποστήριξή σας. Θα ήθελα, συντομία, να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα που θίξατε και εσείς. Πρώτο θέμα, η διαφάνεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Θεωρούμε ότι με την πρότασή μας βρήκαμε μια πολύ καλή ισορροπία. Φυσικά γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα. Και γι' αυτό παρουσιάσαμε ένα θετικό κατάλογο. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο θετικός κατάλογος στηρίζεται στις τρέχουσες πρακτικές, στην ομολογία του ΔΕΚ και στην αξιολόγησή μας για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις περί εμπιστευτικότητας. Οπότε δεν πρόκειται να ευνηδιάσει η πρόταση αυτή τον κλάδο. Επίσης, όταν εκπονήσαμε την πρόταση, διαπιστώσαμε ότι σε αντίθεση με την τρέχουσα πρακτική όπου η ΕΦΣΑ θεσπίζει τους κανόνες με βάση τους οποίους θα λάβει τις αποφάσεις περί εμπιστευτικότητας, τώρα είναι ανοιχτό ο κατάλογος. Οπότε είναι ανοιχτό προς όλους και ο κλάδος το γνωρίζει και η ΕΦΣΑ και η ΜΚΟ και το ευρύ κοινό. Οπότε ως προς την ισορροπία νομίζω ότι έχει βρεθεί χάρη στα στοιχεία αυτού του θετικού καταλόγου. Και εκεί θα πρέπει να δούμε αν μήπω το έχουμε παρατραβήξει. Εμεί πιστεύουμε πάντω ότι έχουμε βρει τη σωστή ισορροπία. Και εδώ δεν μιλούμε μόνο για τα δεδομένα τη αίτηση, αλλά για την αρχή τη προστασία ε, των πνευματικών δικαιωμάτων, τη εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών. Και το ίδιο ισχύει για τι συνεδριάσει που μπορεί να έχουν οι ετούντε με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλεια Τροφίμων κατά την προετοιμασία του φακέλου τους. Σε ό,τι αφορά τους σπόρους και την συμμετοχή των κρατών μέλων, νομίζω ότι υπάρχει μια α, σημαντική καταναλογία αύξηση της ε, συμμετοχής στην ΕΦΣΑ. Είναι αύξηση κατά 80% ε, του προϋπολογισμού, αύξηση του προϋπολογισμού και αύξηση 20 έως 25% του προσωπικού της ΕΦΣΑ. Και όταν συγκρίνουμε την ΕΦΣΑ με άλλους οργανισμούς όπως τον ΕΟΦ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις διαφορές του κλάδου που σχετίζονται με τους οργανισμούς αυτούς ή τα προϊόντα που αξιολογούν ή τον τρόπο λειτουργίας τους. Ο ΕΟΦ ε, εισπράττει κάποια τέλη, ενώ ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων ε, προέρχεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και υπάρχουν διαφορές μεταξύ φαρμάκων και τροφίμων. Είναι αυτονόητο. Όταν παίρνουμε ένα χάπι, ένα φάρμακο, ήδη είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε τους κινδύνους της χρήσης του. Ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε σπαρενέργεια στο μαχόπανο, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα μας βλάψει. Οπότε ε, είναι ένα θέμα που καθορίζει και το βαθμό συμμετοχή του κλάδου στις ε, δράσεις του σχετικού οργανισμού. Είναι σημαντικό πάντως να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ και πιστεύω ότι με τη συμπερίληψη των κρατών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την, το διορισμό εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη, αυτή η ανεξαρτησία διαφυλάσσεται. Επίσης, η ΕΦΣΑ δεν είναι η μοναδική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα κοινό σύστημα όπου θα αναλαμβάνουν ευθύνη και τα κράτη-μέλη. Και θα συμμετέχουν στην όλη συνεργασία. Αυτά ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια αν θέλει να προσθέσει κάτι, αν όχι, πολύ ωραία. Τότε σας ευχαριστούμε άλλους και προχωρούμε με την ημερησία διάταξη. Εν τω μεταξύ, πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, θα ήθελα να καλωσορίσω 24 μέλη από το Ίδρυμα Φίλοι των Ζώων που εκπροσωπούν διάφορες ομάδες και διάφορα πολιτικά κόμματα. Σας ε, καλημερίζω έχουν προσκληθεί από τη συνάδελφο Χάσενκα και βλέπω ότι ζητάει και το λόγο. Παρακαλώ. Ναι. όχι. Μόνο θέλετε να χαιρετήσετε, μάλιστα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας ε, διάταξης. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση εφαρμογής ε, του κανονισμού 1-2005 σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή Αγκρή είχε αναλάβει. της ανατέθηκε μάλλον από τη διάσκεψη των Προέδρων να καταρτήσει αυτή την γνωμοδότηση προκειμένου να διερευνήσει περιπτώσεις κακοδίκησης και παραβιάσεων σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού οι επιτροπές περιβάλλοντος και μεταφορών ε, έχουν διοριστεί ως συνδεδεμένες ε, επιτροπές ε, με μεικτή αρμοδιότητα για όλο το θέμα της εφαρμογής. Φυσικά εδώ συμμετέχει και η δική μας υπηρεσία, κοινοβουλευτική υπηρεσία έρευνας. Αναμένεται να δημοσιεύσει μία δότησε ήδη μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και η κυρία Ραμίρες Βέλα που είναι ε, εκπρόσωπος της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ που έχει έδρα στην Ιρλανδία και ε, από ό,τι γνωρίζω θα υπάρχει και μια αποστολή στην Ιρλανδία από την Επιτροπή μας το Σεπτέμβριο. Είναι εδώ για να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Ντόρμαν, που είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είχα υπογράψει για το να συσταθεί η Δική Επιτροπή για να ερευνήσουμε το θέμα ε, του κανονισμού για την μεταφορά των ζώων. Δεν τα καταφέραμε και είμαι κάπως απογοητευμένος. Τώρα όμως ε, έχω την ευκαιρία να καταρτήσω μία έκθεση εφαρμογής. Ως εισηγητής ανυπομονώ γι' αυτό και είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να αναλάβω αυτό το πολύ σημαντικό καθήκον. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταρτήσουμε μία έκθεση που πράγματι να επικεντρώνεται στο θέμα αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι προφανές ότι ο κανονισμός ε, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τους ε, κανόνες ε, και υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται. Είμαστε στα πρώτα στάδια των εργασιών μας και μας πιέζει ο χρόνος. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια πολιτικά θέματα που θέλω να συμπεριλάβω στην εκθεσή μου και ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε. Θα είναι λοιπόν μια κοινή έκθεση, δική μας έκθεση. Καταρχήν το θέμα ε, της σφαγής ε, στο πιο κοντινό ε, πιο κοντινό σφαγείο έχουμε το θέμα της ε, μεταφοράς ε, των ε, σφάγιων και πρέπει να μεταφέρουμε στο εσωτερικό δίκαιο τους κανόνες. Όμως είναι πολύ διαφορετικό το ποιες κυρώσεις επιβάλλουν οι κυβερνήσεις. Επίσης τώρα το θέμα των εξαγωγών στις τρίτες χώρες. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2015 απεφάνθη ότι ε, κατά τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες ε, πρέπει οι μεταφορείς να σέβονται τους κανόνες ε, και όταν έχουμε μεταφορές στην Τουρκία αυτό αποτελεί πρόβλημα και έχει αναφερθεί συχνά και θέλω να το διερευνήσω. Αλλά έχουμε και που μεταφέρονται στην Κίνα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα σημεία που θα ήθελα να συμπεριλάβω, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που ελπίζω ότι θα κάνουμε είναι ότι θα υπάρχει μια ισχυρή εντολή για την έκθεση αυτή και όπως έχω πει και σε άλλα βήματα, σε άλλα φόρα, ελπίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη πολιτική υποστήριξη από όλες τις ομάδες έτσι ώστε αυτό το σημαντικό θέμα να μπορεί να ξανατεθεί στην ημερήσια διάταξη και να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να μας ακούσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε σχέση με τα ζώα. Αν υπομονώ να ακούσω και τα δικά σας σχόλια. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Γιάννη θέμα. Χάζενκαπ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Σχόλτεμα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μας. Ε, πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι είμαι κτηνοτρόφος. Εμείς τα ε, εκτρέφουμε πάρα πολύ καλά ε, τα ζώα μας. Στις μεταφορές πολλές εταιρείες είναι καλοπροαίρετες, όχι όλες. Και είδαμε και από ντοκιμαντέρ της ε, γερμανικής τηλεόρασης ε, ZDF ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν τηρούνται ούτε στο εσωτερικό της Ένωσης ούτε ε, στις εξαγωγές ζών των ζώων. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η κακομεταχείριση και η βία. Επανειλημμένα εδώ το έχουμε συζητήσει το θέμα και με τον Επίτροπο. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Και τρία-τέσσερα πράγματα έχουν για μένα σημασία που θα ήθελα να τα συμπεριλάβω στην έκθεση και θα κάνω και τροπολογίες. Πρώτον, θα πρέπει να κοιτάξουμε και να ελέγξουμε με ποιο τρόπο η νομοθεσία για τη μεταφορά έρχεται σε σύγκρουση με ε, τη μεταφορά των ζώων. Δηλαδή υπάρχει μια νομοθεσία για τις μεταφορές γενικά και μετά μια διαφορετική νομοθεσία για τις μεταφορές των ζώων που είναι σε σύγκρουση μεταξύ τους και διαμαρτύρονται οι μεταφορικές εταιρείε. και δυσχεραίνεται αυτό. Επίσης για τους χώρους ε, ανάπαυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να μην πω τίποτα χειρότερο στις ε, μεταφορές των ζώων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς πρέπει να βελτιωθεί και πώς μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Ε, είπατε... Ε, ξέρετε ότι οι εμπορικές ε, γραμμές και τα δρομολόγια αλλάζουν. Δεν είναι πάντα στάνταρ. Ε, ανάλογα με τη μέρα, ανάλογα με την ε, ζήτηση και με τις παραγγελίες. Είναι πολύ δυναμικός ο κλάδος και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για τις τρίτες χώρες, νομίζω τα είπα. Και ένα τελευταίο ξανά. Πρέπει να κοιτάξουμε την νομοθεσία για να βελτιώσουμε την εναρμόνιση και να φροντίσουμε να επιβάλλουμε και κυρώσεις. Ισχύουν ένα, αλλά δεν ξέρουμε αν επιβάλλονται οι στα κράτη-μέλη. Και εκεί χρειάζεται εναρμόνιση, γιατί δεν επιτρέπεται οι καλοί μεταφορείς να ε, είναι θύματα αυτής της κατάστασης. Σχόλος, ε, στόχος είναι και η ευζοία και η ευημερία των ζώων και κατά τις μεταφορές. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία και θα πρέπει όλες οι πλευρές να φροντίσουν να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Χάζεκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάθε χρόνο πάνω από 4 εκατομμύρια αγελάδες, 31 εκατομμύρια χείρι, 5 εκατομμύρια πρόβατα, 150.000 ήπι και 1,4 δισεκατομμύρια πουλερικά, κοτόπουλα, χήνες και πάπιες άγονται και φέρονται ανά την Ευρώπη και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και όταν περάσουν ε, τα ευρωπαϊκά σύνορα και πάνε στο εξωτερικό είναι σε πλήρη παρανομία. Ε, με αεροπλάνα, βαπόρια, φορτηγά τα μεταφέρουν ε, με φοβερό καύσωνα και με τρομερό κρύο και κάτι πάει στραβά. Και σκεφτείτε όλα αυτά τα ζώα σε φορτηγά στιβασμένα που περιμένουν ολόκληρες μέρες κάτω από καυτό ήλιο στα εξωτερικά σύνορα. 30.000 κλωσόπουλα πήγαιναν στην ε, Κένια και ε, ε, ψώφισαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις για το πότισμα και δεν ξέρουν πώς να δώσουν στα ζώα να πιούν. Και πολλές φορές έχουμε αγελάδες σε κυοφορία που γεννούν κατά τρεις μεταφορές. Κοιτάξτε τι λένε οι επιθεωρητές από όλες τις οργανώσεις βοήθειας στα ζώα. Αν είμαστε διάφορα ε, ε, σωματεία, ε, ΜΚΟ, ε, φιλοζωικά, που κάνουν τη δουλειά που δεν κάνουν οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν τους αφήνουν. Πραγματικά ε, είναι θλιβερά αυτά τα πράγματα και δεν είναι κάποια επεισόδια. Καθημερινά έχουμε αυτά τα δεινά και την κακοποίηση των ζώων σε διάφορα μέρη, σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Οι άνθρωποι αυτοί εθελοντικά προσφέρουν μια υπηρεσία που δεν κάνουν τα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, εγώ δεν εκπλήσωμαι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεκαετίες ολόκληρες τυφλά επιζητεί το κέρδος και όχι την ευημερία των ζώων. Και κοιτάξτε τι γίνεται στα σφαγεία. Ελέγχουν απλώς τα σφάγια ε, ε, και το προϊόν το κρέας. Αλλά τι γίνεται με τα παραγωγικά ζώα. Γιατί και στα σφαγεία φυσικά ε, με πολύ βίαιο τρόπο και φρικτό ε, θανατώνονται. Έχουμε δει αντίστοιχα σκάνδαλα φρίκης και στο Βέλγιο και στις κάτω χώρες. Δεν θα σταματήσει φυσικά η κακοποίηση των ζώων και τα δεινά αυτά που πρότεινε ο εισηγητής, δεν αρκούν αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει η γεωργία μας, η παραγωγή τροφίμων. Περισσότερες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και λιγότερο κρέας. Και ελπίζω να συμφωνεί και ο εισηγητή. Πάνω από 220 βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη, αριστεροί και δεξιοί, ζήτησαν να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τη μεταφορά των ζώων. Και αυτό ήταν καμπανάκι που δείχνει ότι το Κοινοβούλιο θέλει να εξεταστεί σε βάθος αυτή η φρικτή ε, ε, και ομή πραγματικότητα. Και είμαι απογοητευμένη γιατί κάποιοι υπονομεύουν αυτή την ε, αίτηση και ο πρόεδρος της, Ευρωπαί της Επιτροπής Γεωργίας, ο κ. Σικέρσκι, έπαιξε σημαντικό ρόλο θα πρέπει να στείλει ε, επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ε, μάλλον έστειλε επιστολή και είπε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη Επιτροπή Γεωργία στο θέμα των ζώων. Δεν συμφωνώ μαζί του και εκατομμύρια πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν θέλετε να κάνουμε ακροάσει, δεν θέλετε να κάνουμε ξεχωριστή επιτροπή. Τα, τα διεκπεραιώνουμε αυτά πάρα πολύ γρήγορα και το ξεπερνάμε το θέμα. Δεν ξέρω τι λέει ο Συγητή. Ελπίζω να συμφωνήσει με την Εξεταστική Επιτροπή και να έχει υποστηρίξει και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας. Και τέλος, Πρόεδρε, μια προειδοποίηση. Η σημερινή μου προσκεκλημένη είναι όλοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κόμματος για τα ζώα από διάφορα κράτη-μέλη. Από 11 κράτη-μέλη, για να με ακριβείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνουν αυτά που ζητούν οι πολίτες και τα, ε, ψηφούν τα δικαιώματα των ζώων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι του χρόνου συνάδελφοι, βουλευτές εδώ, για να υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ζώων. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Βλέπω ότι σας υποστηρίζουν και πολύ. Παρακαλώ, συνάδελφε Σράιρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να αντιδράσω αμέσω στα όσα είπε η κυρία Κάζικα ότι και εγώ θα είμαι, ε, και, και εγώ θα είμαι εδώ του χρόνου ε, και άλλοι άνθρωποι που με υποστηρίζουν. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον συνάδελφο Γιάν Χάουτεμα. Περί τίνος πρόκειται. Τι συζητάμε. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν υπερβολές και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν ισχύει μόνο στις μεταφορές των ζών των ζώων αυτό παντού. Ε, ε, ε, ο άνθρωπος παρανομεί και υπάρχουν και μέτρα. Αλλά έτσι όπως αρχίζει σήμερα η συζήτηση νομίζω ότι έχει πάρει πολύ στραβό δρόμο. Και πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει και στην Ολλανδία πώς γίνονται οι μεταφορές. Είναι τέλεια τα φορτηγά και για να πίνουν και για να τρώνε και να ζεσταίνονται και να ψύχονται τα ζώα. Και πηγαίνετε να τα δείτε, είμαι πάρα πολύ περήφανη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε στραβά, ότι όλα πάνε ε, ε, άσχημα. Πάνε μερικά άσχημα, αλλά πάνε και πολλά καλά και θα πρέπει να το ξέρει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το δεύτερο, έλεγχη και χώροι ανάπαυσης. Στην Ολλανδία ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ε, έχω και ιδία πείρα, γιατί είμαι και εγώ κτηνοτρόφος. Όταν δεν υπάρχει έλεγχος εκτινιατρικός, περιμένουν ε, τα φορτηγά να γίνουν έλεγχοι και περνάει μια ώρα και στα σφαγεία δεν υπάρχουν αρκετοί ε, έλεγκτες ε, και επιθεωρητές. Θα πρέπει να τα λέμε και αυτά όταν μιλάμε για ελέγχους. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Εάν λειτουργεί καλύτερα θα φεύγουν και πιο γρήγορα τα ζώα. Και δεν σύμφωνο σε καμία περίπτωση με τον εισηγητή ε, που λέτε να σφάζονται στο κοντινότερο σφαγείο. Είναι οικονομική δραστηριότητα. Εγώ έχω χείρους. Ε, το θέμα είναι ε, ε, πόσο πληρώνει το κάθε σφαγείο. Μπορεί ένα σφαγείο που είναι κοντά μου να μην με πληρώνει αρκετά και ένα άλλο που είναι πιο μακριά 10-15 χιλιόμετρα να πληρώνει περισσότερο και να έχει και καλύτερε συνθήκε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Οικονομική δραστηριότητα είναι. Δεν το λέω για μένα, για όλου του κτηνοτρόφου. Θα πρέπει τα στρεβλά να τα διορθώσουμε, αλλά. Ε, ναι, γελά κιόλα, Άνια. Μπράβο σου. Εγώ δεν γελάω όμω. Γιατί έχω ε, προσωπική πείρα στην ε, εκμετάλλευση ότι θα πρέπει να έρθει ένας ελεγκτής πριν στείλω τα γουρούνια στη Γερμανία και μετά θα έρθει και δεύτερος να ελέγξει τον πρώτο. Αυτά που λέει ο Γιάνν Χάιτεμα ε, ευσταθούν. Ε, μην τα συγχαίουμε όλα και τα ρίχνουμε στο ίδιο τσουβάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος White. White. Ευχαριστώ. Μετά από αυτή την ε, θαυμάσια ομιλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχω πάρα πολλά πολεμοφόδια τώρα για να σας πυροβολήσω κι εγώ και πυρομαχικά. Κοιτάξτε στην Ολλανδία ποιο είναι το πρόβλημα. Για μένα που είμαι αυστριακός αγρότης, ότι εσείς στην Ολλανδία έχετε παραγωγή μαζική, ε, ε, εντατική που εισάγετε ζωοτροφές, δεν έχετε ζωοτροφές, έχετε καλές επιχειρήσεις και τον κύριο Χάρτεμα τον πιστεύω και θέλω να πάω να δω και την εκμετάλλευσή του γιατί σίγουρα θα έχει και κανένα λιβάδι να ταΐζει τα ζώα του αλλά εσείς δεν έχετε λιβάδια και τα εισάγετε ε, από ε, την Αμερική. Εγώ δεν έχω πρόβλημα ότι είναι οικονομική δραστηριότητα και να κάνουμε και business, αλλά όχι στην πλάτη των ζώων για να υποφέρουν τα ζώα. Και σας ερωτώ και προσωπικά, εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας είστε στο πλευρό των κτηνοτρόφων ε, και των γεωργών ή της βιομηχανίας και της μεγάλης business με τα κρέατα. Θέλω να ε, το δω αυτό και θα σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά για να δω σε ποιανού πλευρό βρίσκεστε. Το θέμα δεν είναι η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ως πράσινος θα είχα πολλές προτάσεις για τη βελτίωση ε, του πλαισίου του νομοθετικού για να μεταφέρουμε όσο γίνεται λιγότερα ζώντα ζώα και μόνο εκεί που είναι απολύτω απαραίτητο. Αλλά ποια είναι η έκθεση αυτή. Αν τηρούνται οι νόμοι που ήδη ισχύουν. Και θα πρέπει να ομολογήσω ότι έχετε δίκιο, ναι, για τις μεταφορές των ζώων από τις κάτω χώρες και τη Δανία είναι πολύ καλύτερες ε, πολλές φορές και πολύ πιο κοντά στην νομοθεσία. Ε, έχετε δίκιο, αλλά πιστέψτε με, στην Αυστρία είμαι στο δρόμο με την αστυνομία και σταματώ κάποια φορτηγά που μεταφέρουν ζώντα ζώα και έχω φρίξει με αυτά που βλέπω. Για ελάτε να τα δείτε. 9 στα 10 φορτηγά δεν πληρούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουμε για την Ευρώπη. Και πέρα από αυτό δεν υπάρχει και υποδομή για να τηρηθούν αυτοί οι νόμοι. Χώρια ανάπαυσης, μεταφόρτωσης, ε, δεν υπάρχει υποδομή αλλά δεν υπάρχουν ούτε οι έλεγχοι. Ξέρετε τι θα γίνει αν κάνει ένα καλό ε, έλεγχο ένα κρατήδιο της Αυστρίας, θα κάνουν το γύρο. Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, ξέρω εγώ, για να φτάσουν στην Ιταλία. Θα παρακάμψουν την Αυστρία και οι αστυνομικέ μας αρχές δεν συνεργάζονται. Μπορεί να το κάνουν για την τρομοκρατία, αλλά όχι για τα δυνάτων ζώων. Εκεί τελειώνει η συνεργασία και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το καθήκον πρώτα να φροντίσουμε να τηρούνται οι κείμενοι νόμοι και να ε, γίνεται καλή συνεργασία κατά δεύτερο λόγο ε, στη διασυνοριακή μεταφορά ζών των ζώων. Είμαι σκιώδης ηγητής, θα το παρακολουθήσω το θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ για τις συζητήσεις που θα έχουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφος Κάριν Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείχνει το θέμα πόσο ε, ε, μας ενδιαφέρει και πόσα πάθηκε πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους που υπέγραψαν μια αναφορά, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών που ξεκίνησε ε, ο Νταν Γιόργενσον, παλιός συνάδελφός μας, Stop Tracks λεγόταν, όχι μεταφορές πάνω από 8 ώρες. Βλέπετε λοιπόν πόσο συγκινεί τον κόσμο αυτό το θέμα της προστασίας των ζώων και θέλω να θυμίσω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι τα ζώα είναι ζωντανά πλάσματα που νιώθουν τον πόνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μιλώ τώρα προσωπικά, αλλά προσωπώ τη Μαρία Νόιχελ, την ε, σκιώδη συγκεκριά μας που δυστυχώς σήμερα απουσιάζει. Θα της πω φυσικά ε, τι συζητήθηκε εδώ και με παρακάλεσε να σας παρουσιάσω ε, κάποια σημεία που την ενδιαφέρουν, που ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι για την εφαρμοστική έκθεση τι γίνεται με τις μεταφορές σε τρίτες χώρες. Υπάρχουν κατάφορες παραβιάσεις ε, ε, σε σχέση με την παροχή νερού, ε, τον έλεγχο της θερμοκρασίας κτλ. Εμείς επαγγελματίες ταξιδιώτες είμαστε, καταλαβαίνετε. Φανταστείτε να είσαστε σε ένα βαγόνι που κάνει τρομερή ζέστη, δεν μπορώ να κονηθώ, δεν έχω τίποτα να φάω, δεν έχω τίποτα να πιω. Ή εάν κάθομαι έτσι αναπαυτικά, economy flex και πίνω και κάτι και μπορώ να απλώσω και τα πόδια μου και έχει και κλιματιστικό. Καταλαβαίνετε ε, ότι είναι μεγάλη η διαφορά των συνθήκων. Δεν είναι μόνο πόσες ώρες είσαι καθοδόν, αλλά ποιες συνθήκες επικρατούν στο μεταφορικό μέσο. Δεν αρκούν ε, πάντα ε, οι νομοθεσίες χρειάζονται βελτίωση, αλλά και αυτές που έχουμε είναι καλές, αλλά δεν τηρούνται. Βλέπουμε ότι κάνουν πολλές τάσεις, πολλές μεταφορτώσεις χωρίς ε, χρόνο για την ανάπαυση των ζώων. Και όλο αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το δούμε ξεκομμένο από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναφερθήκαμε στις μεταφορές και πρόσφατα για τις συνθήκες εργασίας των ε, οδηγών φορτηγών συζητούσαμε. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αν έχουμε καλύτερο έλεγχο στις μεταφορές των ζώων, αυτόματα θα έχουμε και καλύτερο έλεγχο ε, ε, σχετικά με την τήρηση των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης για τους οδηγούς, τις οδηγούς των φορτηγών. Κυρώσει Βλέπουμε από την έκθεση ότι σχεδόν είναι ανύπαρκτες, όπως και η έλεγχοι ίσως φραγίζουν ε, την ε, φορτωτική ε, εάν κάνεις αυτές τις παραβιάσεις και θα, θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό και οι επόμενες μεταφορές δεν θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο και μάλλον δεν θα περνάνε από αυτά τα μέρη όπου γίνονται αυτοί οι έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζονται όλα αυτά για τη μεταφορά μέχρι τη σφαγή την ίδια, αλλά ε, ε, χωράει και μεγάλη βελτίωση, όπως λέει και η έκθεση. Και σίγουρα θα πρέπει να προτιμούμε τη μεταφορά κρέατος και όχι τη μεταφορά ζών των ζώων. Ε, Χθε μιλούσαμε συνέχεια για την προσέγγιση ενία υγεία, One Health και γενικά για την ευημερία των ζώων θα πρέπει να προσέχουμε ότι ακόμα και αν πηγαίνουν στη σφαγή θα πρέπει τα ζώα αυτά να μεταφέρονται με τις καλύτερες γενικές, ε, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Γιατί όταν το ζώο υποφέρει κατά τη μεταφορά, υδρώνει και τα λοιπά, εκρίνονται και διάφορες ε, ουσίες και τοξίνες που περνούν στο κρέας και είναι κακό για την ανθρώπινη υγεία έξω και το One Health. Ξέρω ότι έχει αρμοδιότητες και η Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι θέλουμε να πιέσουμε ε, και στα προϊόντα, κατεργασμένα προϊόντα που περιέχουν κρέας, όχι στο ίδιο το κρέας, να γίνεται σωστά η επισήμανση και να βλέπουν στην ετικέτα οι καταναλωτές από πού προέρχεται το κρέας που έχουν στο μαγειρεμένο προϊόν που αγοράζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κάριν. Ωραία. Ακούσαμε όλους τους συναδέλφους που είχαν ζητήσει το λόγο. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, ε, Ραμίρες Βίλα, από την Δέλτα ΣΑΝΤΕ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Για την ευκαιρία που μας ε, δίνει να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Εμείς χαιρετίζουμε την έκθεση και περιμένουμε με ανυπομονησία την έκβαση. Στο θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων, στη μεταφορά, αυτό είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρόνια ολόκληρα και γι' αυτό εκφράζουμε την αμέριστη ε, διάθεσή μας για συνεργασία με την Επιτροπή για να δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται. Όντως είναι περίπλοκο το θέμα, αφορά πολλά είδη, πολλά υπουργεία μεταφοράς και έχει και μια διεθνή διάσταση. Ένα από τα προβλήματα είναι τα αξιόπιστα στοιχεία που δύσκολα συγκεντρώνουμε. Έχουμε επίγνωση κάποιων προβλημάτων κατά την εφαρμογή του κανονισμού, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο να προσδιορίσουμε την σχετική σημασία ή τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων. Έχουμε επίγνωση των, προγραμμάτων με, των προβλημάτων μεν, αλλά δεν γνωρίζουμε τις διαστάσεις των συνεπειών ή το εύρος των προβλημάτων μη συμμόρφωσης. Κάποιες πληροφορίες τώρα για, το, για τις τρέχουσες προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το μελλοντικό έργο για τον κανονισμό. Την τελευταία διετία είχαμε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη μεταφορά ζώων προς εξαγωγές ε, στις ε, ε, τρίτες χώρες, ιδιαίτερα την Τουρκία. Έχουμε πραγματοποιήσει επισκέψεις στην Τουρκία, τη Βουλγαρία και άλλα κρατημέλη και προετοιμάζουμε τη σχετική έκθεση για τέτοιου είδους μεταφορά. Θα τη δημοσιεύσουμε εντός διμήνου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει επίσης και ένα έργο για τα livestock vessels Σκάφη. Τα πλοία που μεταφέρουν ε, ε, ζώα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές, ε, τα στοιχεία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει θετική τάση υπέρ της εφαρμογής του κανονισμού. Επίσης, διαπιστώνεται υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των μεταφορέων κατά την άφηξή του στα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε με τα κράτη-μέλη τα τελευταία 5-6 χρόνια μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη μεταφορά των ζώων και χάρη σε αυτό το δίκτυο έχουμε εκπονήσει πολύ σημαντικά έγγραφα που μπορεί να μην έχουν νομική ισχύ αλλά πραγματικά συμβάλλουν στην εναρμόνιση της εφαρμογής και στην ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε για παράδειγμα έγγραφο για τη μεταφορά πουλερικών που συμφωνήσαμε με τον κλάδο των πτυνοτρόφων και ένα έγγραφο κοινό που συμφώνησαν τα κράτη-μέλη για τα πλοία που μεταφέρουν ε, ζώα και έχουμε και άλλα έγγραφα. Επίση, τον περασμένο Νοέμβριο συστήσαμε μια υποομάδα για τη μεταφορά ζώων στα πλαίσια τη πλατφόρμα ε, για την ευζοία. Και μάλιστα ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η υποομάδα τη εργασία τη ε, και ε, θα επικεντρωθεί σε τρει τομεί. Και πριν τα τέλη του 2019 θα υποβάλει σχετική μελέτη. Τα τρία θέματα είναι η εξαγωγή βοηδών, υπερβολικές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά και μεταφορά των ζώων. Επίσης, θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες μεταφοράς ε, προς τις τρίτες χώρες για πολλά είδη, ε, χειρούς, εγωπρόβατα, άλογα και ούτω καθεξής. Και θα έχουμε και μια φάση ε, για την διάδοση αυτών των εγγράφων μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασής τους σε πολλές γλώσσες. Όπως είπα, χαιρετίζουμε την έκθεση. Δεν θέλουμε τώρα να εμπλακούμε στη συζήτηση για το κατά πόσο μεταφορά σε μεγάλη απόσταση θα πρέπει να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται. Έχουμε νομοθεσία που επιτρέπει τη μεταφορά των ζώων και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να κρίνουμε αν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο, ποια είναι τα ωφέλη ή τι γεωργικό μοντέλο ή κτηνοτροφικό μοντέλο θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό το παρόντος, ούτε δική μου αρμοδιότητα. Και σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφος θέλει το λόγο, ναι να προσθέσω μια επικοδομητική πρόταση. Θέλω να επενθυμίσω στους συναδέλφους αλλά και στην Κομισιόν ότι ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ένα δημοσιονομικό τέτοιο πρόγραμμα ε, για τα σφαγεία. Μιλήσαμε και με την, το συζητήσαμε με την ομάδα για την ευημερία των ζώων ε, και θα ήθελα να υποστηρίξετε την πρόταση αυτή για τα κινητά σφαγεία και θα θέλαμε, παραδείγματο χάρη, να έχουμε κινητά σφαγεία που να είναι πιο κοντά στι εκμεταλλεύσει και ίσως ε, να συνεισφέρουν σε ένα μέρος της λύσης ε, στο να μειωθούν ε, οι μεταφορέ ή τουλάχιστον οι μακρινές μεταφορές των ζώων. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλήσω να υποστηρίξετε την πρόταση αυτή. Πολύ ωραία. Τώρα ο εισηγητής για τις καταληκτικές του παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η πρώτη συζήτηση μας δείχνει ότι ήδη συμφωνούμε σε πολλά σημεία και στο ότι, ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τη μεταφορά των ζώων. Έχουμε διαφοροποιημένες καταστάσεις στις διάφορες χώρες. Πρέπει να δούμε πώς οι χώρες αυτές θα εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνες. Όταν μιλάμε για τους ελέγχους ε, κατά τη φόρτωση των ζώων πριν από τη μεταφορά, είναι διαφορετική και επίσης διαφέρουν και οι κυρώσει στη Δανία, παραδείγματος χάρη. Θα μπορεί να επιβληθεί ε, κάποιο πρόστιμο στον ε, μεταφορέα επειδή δεν έχει μεταχειριστεί καλά τα ζώα. Υπάρχει λοιπόν ένας ε, κίνδυνος αν στέλνει κανείς ζώα για μεταφορά τα οποία δεν είναι καλά στην υγεία τους. Θέλουμε να σταματήσουμε τέτοιες πρακτικές. Εμείς προτείνουμε να σφαγιάζουμε τα ζώα αν έχουν μεταφερθεί για σφαγή. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να μεταφέρουμε άλογα για σφαγή στην Ιταλία παραδείγματο χάρη θα μπορούσαμε να τα θανατώνουμε στην ε, Δανία και θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα καταψυγμένα ε, σφάγια στην Ιταλία για περαιτέρω επεξεργασία. Όμως ε, θα πρέπει να δούμε το θέμα της νομοθεσίας. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της νομοθεσίας για τις μεταφορές και της νομοθεσίας για τις μεταφορές των ζώων. Εγώ νομίζω ότι κάθε χώρα θα πρέπει να υποχρεούται να διασφαλίζει το σεβασμό Τη νομοθεσία. Ε, δεν πρέπει να το πετούμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τα κράτη-μέλη. Επίση, νομίζω ότι όσοι επιλέγουν ε, διαδρομέ ε, μέσω χωρών που ξέρουν ότι δεν υπάρχει έλεγχη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα βελτιώσουμε τις συνθήκες για τα ζώα, πρόσβαση στο νερό, παραδείγματο χάρη, ή παραδείγματο χάρη ένας χώρος ε, ε, για τους χείρους ε, που να μπορούν να παίξουν, κάτι που να δείχνει ε, παραδείγματο χάρη ότι μπορούν να έχουν δικαιώματα, ε, να μπορούν ε, παραδείγματο χάρη να κάνουν και ένα μπάνιο τα ζώα. Επίσης, αν υπάρχουν πολύ ψηλέ θερμοκρασίες χωρίς πρόσβαση στο νερό, αυτό είναι απαράδεκτο. Στο Στρασβούργο την τελευταία φορά άκουσα ότι σταμάτησε το τρένο και δεν είχαν πρόσβαση στο νερό οι ταξιδιώτες. Ξέρετε, αν ήταν ε, χείροι θα είχαν πρόσβαση στο νερό όμως. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό μας δείχνει ότι έχουμε ένα project. Συμφωνούμε βέβαια στο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε πόσο μπορούμε να πιέσουμε σήμερα. Επίσης, και εγώ υπέγραψα για να έχουμε μια εξεταστική επιτροπή, όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας για να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες για τα ζώα. Αυτό δεν θα σταματήσει λόγω των εκλογών, θα συνεχίσει και στην επόμενη θητεία. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους και την ε, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα, γιατί θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημέρας της διάταξης, που είναι η παρουσίαση από ε, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης ε, Άγκρη. Θα έχουμε μια παρουσίαση για διάφορα εμπορικά ζητήματα με γεωργική διάσταση. Αυτό αφορά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Για αυτή τη ε, συνεδρίαση θα συνεδριάσουμε και κλεισμένων των θυρών. Έτσι λοιπόν, ας κάνουμε 2-3 λεπτά διάλειμμα και να ζητήσουμε στους βοηθούς και στους υπολείπους να εγκαταλείψουν την αίθουσα.